Συνάδελφοι, σύμφωνα με τριμερήσια διάταξη πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή των κοσμητόρων του Κοινοβουλίου. Έλαβα τις εξής υποψηφιότητες. Ο κύριος Γκέριγκερ, η κυρία Γκέριγκερ, ο κύριος Χίγκινς, η κυρία Λούλινγκ, ο κύριος Μαστάλκα, ο κύριος Νιούτον Ντάν, ο κύριος Νίκολσον, η κυρία Όμενε Ρόιτεν και ο κύριος Σπερόνι. Οι υποψήφοι με ενημέρωσαν ότι δέχονται τις αντίστοιχες ε, υποψηφιότητες και εφόσον τον νου, ο αριθμός των υποψηφιότητων ξεπερνά τον αριθμό των εδρών που θα πρέπει να ε, καλυφθούν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία μυστική ψηφοφορία. Όποτε και θα πράξουμε, θυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού αυτές οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για την εκλογή των αντιπροέδρων. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν στην εκλογή με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να μπορέσουμε όλοι να εξοικειωθούμε με το ηλεκτρονικό σύστημα, και κυρίως για όσους είναι νέοι εδώ, νεοεκλεγέντες, θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε ήδη στα έδρανά σας ένα ενημερωτικό ε, δελτίο για την χρήση των καρτών που έχετε, αλλά νομίζω πως είναι χρήσιμο να θυμίσουμε κάποια σημεία. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε στη σχισμή την κατάλληλη την κάρτα με το ηλεκτρονικό μικροτσίπ προς τα κάτω. Σε περίπτωση λάθος θα υπάρξουν βοηθητικές οδηγίες στην οθόνη που έχετε μπροστά σας. Επίσης υπάρχουν οι εξής πληροφορίες στην οθόνη. Ο αριθμός της κάρτας ψηφοφορίας, το όνομα του βουλευτή και η ημερομηνία. Τρίτο σημείο. Μετά την ανακοίνωση του καταλόγου των υποψηφίων και την έναρξη ψηφοφορία, στην οθόνη σας θα εμφανιστούν οι εξής πληροφορίες. Το αντικείμενο της ψηφοφορίας, ο κατάλογος των ε, υποψηφίων και ο αριθμός των εδρών που θα πρέπει να καλυφθούν. Τέταρτο σημείο, θα πρέπει να τοποθετηθείτε για τον όνομα του προεπιλεγμένου υποψηφίου πιέζοντας ε, τα μπλε κλίκτρα προς το κάτω ή προς τα πάνω και να εκφράσετε έτσι την ψήφο σας ε, πιέζοντας ε, το πλήκτρο συν που είναι στα αριστερά της ε, κονσόλας σας. Θα ανάψει το μπλε φωτάκι και ένας αστερίσκος θα φανεί δίπλα στο όνομα. Τώρα, για να σεβαστούμε την μυστικότητα της ψηφοφορίας, η μετακίνηση του Κέρσορα καταργεί τον αστερίσκο, ε, τον διαγράφει δηλαδή. Για να δούμε το υπόλοιπο του καταλόγου θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον κέρσορα μετά το τελευταίο όνομα που υπάρχει στην οθόνη και τότε θα φανούν και τα υπόλοιπα ονόματα. Αν θέλετε να εκφράσετε την ε, παρουσία σας ε, στις εκλογές χωρίς να ψηφίσετε για κάποιον υποψήφιο μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 0 που είναι το κεντρικό πριν από την ανακοίνωση του τέλους της ψηφοφορίας είναι δυνατόν να αλλάξει κανείς ε, την επιλογή του τοποθετώντας ε, άλλο όνομα και πιέζοντας ε, το πλήκτρο 0 ώστε να ακυρώσει την θετική του ψήφου, να τοποθετηθεί έπειτα με τον κέρσορα στο όνομα ενός άλλου υποψήφιου και να πιέσει το πλήκτρο συν. Τέλος, για να δείτε όλους τους υποψηφίους που έχετε ψηφίσει, να πιέσετε το πλήκτρο χ κάτω από την οθόνη στα αριστερά. Αν το πιέσετε μια δεύτερη φορά θα ε, ακυρωθούν οι αστερίσκοι. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Με συγχωρείτε που μιλάω λίγο δασκαλιστικά. κυρίως για τους νέους ε, βουλευτές. Ας κάνουμε λοιπόν μια επιλογή. Ας διαλέξει ο καθένας δυο ε, υποψηφίους από τους έξι που προτείνονται στον εξή κατάλογο. Φυσικά, ο πρώτος είναι ένας περίφημος ε, ε, τραγουδιστής, είναι όλοι τραγουδιστές, που δυστυχώς χάθηκε. Δεύτερος τενόρος είναι ο Πλάσιντο Ντομίνγκο, τρίτος είναι ο Ζωζέ Καρέρας και μετά έχουμε τρεις σοπράνο, την Τζούλια Μιγένες, την Μοσεράτ Καμπαγέ και την Τζέσι Νόρμαν. Λοιπόν, επιλέξτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Io non να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 Θυμίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο δύο από τους υποψήφιους. Dei cinque candidati. L'onorevole Silvestri. No, sì. No, no, no. L'apparecchio che non funziona. Sì, ho già, ho già chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz. Ορίστε κύριε Σούλτ, Πρόεδρε, πρόεδρε, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να εξηγήσετε κάτι. Αυτό είναι δοκιμαστική ψηφοφορία. Στη δοκιμαστική μπορεί να ψηφίσει κανεί μόνο δύο. Τον Παραγιώτη και Παβαρότη και την άλλη, πώς τη λένε, Μοσεράτ Καμπαγιέ. Μετά στους κοσμήτορε όμως, πέντε θα ψηφίσουμε. Έτσι, να τα ξέρουμε αυτά τώρα στο τεστ μόνο δύο, για να μην μπερδευόμαστε. Πολλοί συνάδελφοι έχουν οδηγηθεί σε σύγχυση. Στη δοκιμαστική δύο, στην κανονική πέντε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σούλτς. Σας ευχαριστώ που προτρέξατε τον όσον θα έλεγα πριν από την επόμενη ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ για το ζήλο που δείχνετε. Ψηφίσατε όλοι? Ο κύριος, κυρία Σιλβέστρη που δεν ψήφισε. Κύριος, ε, πρόεδρε, καταρχήν. Σας ευχαριστώ που βάλατε τον Παβαρότη πρώτο, αλλά να πω και κάτι άλλο. Αφού έχουμε βάλει εκείνους τους τάδε δύο που θέλουμε να ψηφίσουμε, πρέπει να επικυρώσουμε την ψήφο μας ή πρέπει να μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται επικύρωση. Άρα βάζουμε ένα αρχή μπροστά και τέλο.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 Λοιπόν, αρκεί. Αρκεί η δοκιμή θα έλεγα. Δεν έχει κανένα νόημα. Όσο προ την εκλογή των κοσμητών, λοιπόν, τέλο τη ψηφοφορία. Sì. I Posso annunciare il Λοιπόν, για να δούμε. Λουτσιάνο Παβαρότη, 380 ψήφοι. Ντομίνγκο Πλάσιντο, 283. Ζωζέ Καρέρα, 213. Καμπαγέ Μοσερά, 178. Τζέσι Νόρμαν, 117. Μιγγέλες Τζόνσον Τζούλιον, 109. Αυτά. Αυτή ήταν η δοκιμή. C'è una richiesta di, di parola dell'onorevole prego. Ο κύριο Κασίνη παρακαλώ. Δεν ξέρω αν καταλάβαν όλοι την προφορική επεξήγηση της ψήφου, της ψηφοφορίας. Παρακαλώ, να εξηγήσετε ακόμα μια φορά πώ ψηφίζουμε. Io non lo Ε, δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται ξανά μανά τα ίδια. Εξάλλου τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δείχνουν ότι η ταχύτης ε, απορρόφησης ε, των νέων γνώσεων είναι τεράστια. Allora, procediamo alla elezione vera. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην πραγματική ψηφοφορία των κοσμητόρων να επαναλάβω τα όσα δήλωσε ο κύριος Σούλτς, ότι πρέπει να εκλεγούν πέντε συνάδελφοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέντε.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 Ωραία, λοιπόν, μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Ε,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 Ψήφισαν 696. Άκυρα 2. Άρα έχουμε 694 ψηφίσαντες, η πλειοψηφία είναι 348, η απόλυτη πλειοψηφία. Γκέριγκερ 398, Higgins 352, Λούλινγκ 322, Μαστάλκα 206, Νίκολσον 174, Νιούτον 171, Όμεν 161, Σπερόνι 145. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα εκλέγεται με τον πρώτο γύρο, εκλέγονται με τον πρώτο γύρο οι κύριοι Γκέριγκερ και Χίγκινς, τους οποίους συγχαίρω και συγχαίρουμε όλοι. Restano dunque da assegnare altri tre seggi ed è Πρέπει να πληρωθούν άλλες τρεις θέσεις. Πάμε στο δεύτερο γύρο λοιπόν ψηφοφορίας. Εκεί όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ πως διατηρούνται οι υποψηφιότητες του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας. Ε, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από ό,τι βλέπω. Ωραία. Δεύτερος γύρος θα γίνει στις 3. Μα συνάδελφοι, εγώ το έκανα για να, την υγεία σα για το ποσοστό υπογλυκαιμία. <laughs> Αλλά δεν έχετε προβλήματα υγεία, συμφωνώ να ψηφίσουμε αμέσω να τελειώνουμε. Dobbiamo soltanto dare il tempo eh, per la Μόνο λίγο χρόνο για να μπουν τα ονόματα στον υπολογιστή, να φύγουν αυτοί που ήδη έχουν εκλεγεί. avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti Ωραία, λοιπόν, έχουν μειωθεί οι υποψήφοι τώρα και ο αριθμός των ε, ψήφων είναι τρεις. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει τρεις υποψηφίους τώρα. Όχι πέντε, τρεις.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 ancora problemi con i dispositivi? Tutto bene? Possiamo chiudere la votazione? Possiamo chiudere la votazione? Μπορούμε να κλείσουμε την ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Allora, la votazione... Ωραία, τέλος της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Εψήφισαν 699. Δύο άκυρα. Άρα 697 ψήφοι, πλειοψηφία 3, 4, 9, 349. Η κυρία Λούλινγκ, 327, Μαστάλκα, 2, 283, Νιούτον Ντάν, 202, Όμεν Ρόιτεν, 187, Νίκολσον, 172, Σπερόνι 130. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταφύγουμε στον τρίτο γύρο. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προχωράμε στην τρίτη ψηφοφόρια. Ισχύει απλή πλειοψηφία. Όπως και για τους αντιπροέδρους. Δεν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 Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Hanno votato tutti? Possiamo chiudere la votazione? Ψηφίσατε όλοι να κλείσουμε την ψηφοφορία. Ωραία, ευχαριστώ. Τέλος της ψηφοφορίας λοιπόν. Hanno votato 7 Εψήφισαν 705. Δύο άκυρα. 703 έγκυρη. 306 ψήφους η κυρία Λούλινγκ. Ο Μαστάλκα 293. Νιούτον Ντάν 208. Όμεν Ρόιτεν 186. Νίκολσον 176. Σπερώνη 131. Άρα λοιπόν εκλέγονται ως κοσμήτορες οι κύριοι Λούλινγκ, Μάσταλκα, Νιούτον Ντάν τους οποίους συγχαίρουμε. Σας παρακαλώ να μην φύγετε από την αίθουσα γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλη μια ψηφοφορία. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση της πρότασης για την αριθμητική σύσταση των επιτροπών. Σημαντική ψηφοφορία μάλλον. Πριν από αυτήν θα ήθελα να ανακοινώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον, ε, τη σειρά με την οποία εκλέγησαν. Η σύσταση λοιπόν του Προεδρείου θα τροποποιηθεί ε, σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι η αριθμητική σύσταση των μόνιμων επιτροπών. Σύνθεση, συγγνώμη. Έχουμε την πρώτη τροπολογία που έχει υποβληθεί από την ομάδα Ελευθερία και Δημοκρατία και άρα ψηφίζουμε την τροπολογία ε, την νούμερο 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγώ χρειάζομαι γυαλιά, αλλά και χωρίς τα γυαλιά μπορώ να δω πώ υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία κατά αυτή της τροπολογίας. Άρα λοιπόν απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, κανείς δεν απέχει. Οπότε, το ψήφισμα εγκρίνεται. Ευχαριστώ τους συνάδελφους και τις συναδέλφους. Ε, διακόπτεται η συνεδρία. Θα ξαναρχίσουμε στις 3. Καλή όρεξη σε όλους. Το αξίζεται. Να φάτε καλά.